Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ε, χαιρετήσω στα θεωρία των επισκεπτών την αντιπροσωπεία μας από το Κογκρέσιο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Συμπρόεδρο στην Μεκτή ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή, τον κύριο Κλειφ Στέρνς και τους επτά συναδέλφους που τον συνοδεύουν. Καλώς ήρθατε και χαίρομαστε πολύ που σας βλέπουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συνάδελφοι από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται εδώ ε, για, την, συμμετοχή στον διάλογο, τον διατλαντικό κοινοβουλευτικό διάλογο στην Κοπενχάγη το Σάββατο και την Κυριακή μαζί με τους συναδέλφους από τις ΗΠΑ θα ε, ξέρετε ασφαλώς ότι είχαμε την ε, συνεδρίαση αυτή και θα λάβουν σήμερα μέρος στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής των Εξωτερικών ολοκληρώνοντας έτσι τις εργασίες τους εδώ. Οι αρχές της Γαλλίας με ενημέρωσαν για την εκλογή των εξής κυρίων, κυρίων και κυρίων από 16 Μαου 2012, Ερίκ Αντριού που αντικαθιστά τον κύριο Καντέρα Ρίφ, τον κύριο Ζων Ζακόμπ Μπισέπ που αντικαθιστά τον κύριο Πασκάλ Κομφέ,